ο κόσμος να, ε, να, να, να, να, να, να αμείβεται για τις προσπάθειές του, για τη δημιουργία του, αλλά ταυτόχρονα προστατεύονται και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Γι' αυτό θα μας προσχωρήσει και στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Τέλος της συζήτησης, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση του Ζεβάν Λαβία, προπολογισμό 2013, εντολή για τον τριμερή διάλογο και δίνω αμέσως το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή Τζοβάνι Λαβία. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η ψηφοφορία για την εντολή για το τριμερή διάλογο ε, γίνεται σήμερα ε, σε μια κρίσιμη φάση για την Ευρώπη, αλλά κυρίως κρίσιμη φάση για την αυριανή Ευρώπη. Το Συμβούλιο της 28-29 Ιουνίου αποφάσισε να ελαβει ένα, μια σειρά μέτρων για να εγγυηθεί μια οικονομικά σταθερή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί παρά να χαροποιήσει, γιατί οι αρχηγοί των κυβερνήσεων έδειξαν ως ε, μια διέξοδο ε, από την κρίση αυτά που εμείς από την αρχή της κρίσης λέγαμε υποστήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης κυρίως για τους νέους και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που εμείς είχαμε θέσει ως Κοινοβούλιο γνωρίζοντας την άμεση ανάγκη ανάκαμψης της οικονομίας μας που δεν μπορεί παρά να γίνει μέσω μιας ανταγωνιστικής ανάπτυξης μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα που θα εγγυάται στήριξη των νέων για να μπουν στην αγορά εργασίας. Έπειτα υπάρχει ανάγκη μιας επαρκ... ενός επαρκούς επίπεδου πληρωμών για να εγγυηθούμε τις δαπάνες που προκύπτουν από τα διάφορα προγράμματα, κυρίως στις κατηγορίες 1α, 1β και 2. Όπως γνωρίζουμε αυτό είναι ένα από τα κεντρικά θέματα των διαπραγματεύσεων. Είναι στο πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν διαφορετικοί προσανατολισμοί όπως έχουμε δει μέχρι σήμερα από ορισμένα κράτη-μέλη. Θα ήθελα ωστόσο να θυμίσω ένα σημείο στα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην αυριανή ψηφοφορία μέσω μιας προφορικής τροπολογίας όπου το Συμβούλιο επιβεώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ξαναφέρει την Ευρώπη σε ένα δρόμο εφιούς, βιώσιμης και καθολικής ανάπτυξης. Πιστεύω πως ε, μια τέτοια ένδειξη πολιτικής βούλησης δεν μπορεί μετά να μην ακολουθηθεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς όλων των κρατών μελών, ώστε να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να ε, μπορέσουν να επιτύχουν τους ε, στόχους. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω πως ε, οι υποχρεώσεις πληρωμών που προτείνεται από την Κομισιόν στο σχέδιο προπολογισμού βασίζονται σε εκτιμήσεις που έχουν γίνει από τα ίδια τα κρατημέλη, μελη τις έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω η Κομισιόν και έπειτα τα κρατημέλη θα πρέπει να τηρήσουν όσον αφορά τα ΡΑΛ και την ε, διαθεσμική συνάντηση για τις πληρωμές που έγινε στις 30 Μαΐου θα πρέπει να προσθέσω ότι θεωρώ βασικό για τη σωστή εξέλιξη διαδικασία τη φετινή και για την επιτύχηση ενός αποτελέσματος που θα βασίζεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών μια διαρκή άσκηση παρακολούθησης των δαπανών, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε λογαριασμό, να, να συνειδητοποιούμε μάλλον τις ανάγκες, τις μελλοντικέ και γι' αυτό χρειάζεται στενή οργανική συνεργασία που δυστυχώς δεν υπήρξε. Έπειτα θα πρέπει να αποφύγουμε τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της περσινής διαδικασίας, ε, δηλαδή να, και, που οδήγησαν στη διορθωτικό προπολογισμό για τις πληρωμές μέσα στο 2012. Αν λάβουμε υπόψη το 2013 είναι η τελευταία χρονιά για τις δημοσιονομικές προοπτικές και ότι περιμένουμε αύξηση του επίπεδου των πληρωμών θα πρέπει να αποφύγουμε μια επικίνδυνη διολίσθηση των πληρωμών από το 2012 προς το 2013. δεν υπάρχουν όμως μόνο οι πληρωμές, αλλά και ανάγκη ενός επαρκούς επίπεδου ανάληψης υποχρεώσεων, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια φάση κρίσης, όπως το είπε και το Συμβούλιο, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη. Και γι' αυτό, στο επίπεδο των υποχρεώσεων, Χρειάζεται να δώσουμε ισχύ στις πολιτικές μας προτεραιότητε και να προωθήσουμε τι απαραίτητε επενδύσεις για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση για να βγούμε από την κρίση. Τελευταία πτυχή που είναι σίγουρα σημαντική και σχετίζεται με τη χρηματοδότηση Twitter. Ήδη Έχουμε σημειώσει την πρόταση της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει κάποιους πόρους που έχει πάρει μέσω της περικοπής ε, του 7ου του πλαισίου και να επαναλάβουμε ότι το Κοινοβούλιο στο σκοπεύει, όπως ε, εξάλλου έχουμε πει στην κοινή δήλωση, ε, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του μέσα στο πλαίσιο της, του δημοσιονομικού κανονισμού και της Διοργανική συμφωνίας. Θα κλείσω ευχαριστώντας του συναδέλφους και κυρίως τους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Και στρεφόμενο ε, προ τον ε, Πίστροπο Λεβαντόφσκι, αφού λείπει εκπρόσωπο του Συμβουλίου, να τον καλέσω για στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια όλες τις διαδικασίες που ελπίζω πω θα ολοκληρωθεί με επιτυχία με τους κατάλληλους, ε, τα κατάλληλα κονδύλια και εντό των προθεσμιών που προβλέπει η συνθήκη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Έχουμε εδώ δύο παράλληλες διαδικασίες ως συνήθως επί τη βάση της πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 για αυτό το σχέδιο προπολογισμού και αυτό γίνεται μέσα στη σημερινή συγκεκριμένη συγκυρία. Θεωρείται η δημοσιονομική εξυγίανση ως η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Όμως από την άλλη μεριά, ακόμη και σε καιρούς κρίση χρειάζονται οι επενδύσεις και επομένως έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και απασχολή στο μέλλον και αυτά τα είπαμε ει τα συμπεράσματα της τελευταίας ε, συνάντησης κορυφη Νομίζω ότι για την απάντηση την έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το σχέδιο του πρόγραμμα του 2013. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σωστά και τότε ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο... Είχαμε δει τότε ότι ο κύριος Λαβία πήγαινε στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να γίνουν οικονομίες, εξοικονομίες δαπανών και θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε μόνο 2% ε, πιστώσεις υποχρεώσεων αλλά είπαμε ότι η άλλη μεριά θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για ό,τι έχουμε δεσμευθεί και νομικά μέχρι το 2013. Οι μεσονομικές προοπτικές ε, δεν θα πρέπει να εκπλήσουν κανένα γιατί στο τέλος της περίοδου των προοπτικών κάποια προγράμματα θα φτάσουν περίοδο οριμότητος και οι πληρωμές τότε θα επιταχυνθούν σε ρυθμό. Επίσης αυτό αφορά και τη χρήση του 2013, οπότε και το νη συν 1, νη συν 3 σημαίνει ότι εμείς θα πληρώσουμε το 2013 το αργότερο τις υποχρεώσεις από το 2011 και 2012. Τώρα, όσον αφορά τι πιστώσει πληρωμών, πρόκειται περί συλλογική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα μόνο δικό μα. Και είδαμε επομένω ε, τι γίνεται όσον αφορά όλε εκείνε τι περιοχέ που έχουν δυνατότητε ανάπτυξη, ε, του στόχου τη συνοχή, γιατί η αναβολή των πληρωμών δεν είναι λύση. Ε, γιατί τότε έχουμε πρόβλημα ρευστότητα στα κράτη-μέλη. Ή από την άλλη μεριά έχουμε απλώ ε, περικοπή των δυνατοτήτων περιπτώσεων ε, επενδύσεων και αυτό είναι ε, κίνδυνος για το μέλλον. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβετε υπόψη και όσα είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Προπολογισμών στο Κοινοβούλιο να το λάβετε απόψη αυτό και στο μέλλον σε σχέση με τα επίπεδα των πληρωμών τέλη Μαΐου. Νομίζω ότι υπάρχει ο και περισσότερη κατανόηση για το τι θα γίνει όσον αφορά την, το, το πολιετές ε, πλαίσιο, χρηματοδοτικό πλαίσιο όπως τα είπε ο κύριος ε, Λαβία ε, πολλές φορές αγνοούμε το τι θα χρειαστεί το 2013 και πολλές φορές τίνει το Συμβούλιο να θέλει να επιβάλλει περικοπές. Όμως από την άλλη μεριά καταλάβετε ότι οι περικοπές δεν προέρχονται από εμά, έρχονται από τα κράτη-μέλη. Εμεί είμαστε πιο απεσιόδοξοι από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το επίπεδο πληρωμών για το 2013. Παρ' όλα αυτά ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει συνεργασία στα κέντρα των αποφάσεων, στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ τον, τον που μας έκανε τώρα και αυτή την, την, ε, τη λίστα με τις ε, τα βασικά προγράμματα, τι προτεραιότητε, είναι τα πράγματα πιο εύκολα του 2013 και για άλλη μια φορά. Επομένω, εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξο ότι ακόμα και με τι ε, σημερινέ τόσο δύσκολε συνθήκε θα μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή λύση για τον προπολισμό τη επόμενη κρίση. Grazie Commissario. La parola per la Commissione Affari Esteri all'onorevole Εξ ονόματος Επιτροπής Εξωτερικών, η κυρία Γιατρεμάκη. Ευχαριστώ. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει οικονομίες στα πλαίσια της κρίσεως και ε, βλέπω ότι προτίθεται μία αύξηση του προπολογισμού κατά 7% πράγμα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα χρέη των εθνικών προϋπολογισμών και είναι το ίδιο ποσό το οποίο περιεκόπη από τον προπολογισμό για την υγεία στη χώρα μου για τον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων ε, προβλέπεται μία αύξηση 7,5% παρόλο που ε, επιδεινώνεται η κατάσταση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Συγχρόνως όμως η, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπεύθυνοι για την εξωτερική ε, πολιτική λέγουν ότι η κατάσταση είναι σταθερή. Ε, ε, το μήνυμα πρέπει να είναι ενιαίο, ότι πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσεις πόρων, αλλά πρέπει το περιβάλλον όπου εργάζεται κανείς να είναι ασφαλές. Εάν δηλαδή τα κράτη-μέλη κάνουν οικονομίες, πρέπει να εξοικονομήσουν χρήματα χρήματα και ε, εις ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μίτσελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τζοβάν Λαβία για την πολύ εντατική δουλειά που έκανε εδώ. Στον χρόνο που έχω να πω ότι καταλαβαίνω πως ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να θέλουν να μειώσουν τη συμβολή τους προς την αναπτυξιακή βοήθεια σε αυτούς τους πολύ δύσκολου καιρού. Αλλά το 0,7% καταβάλλεται στο GNI. Άμα το, το, το ΑΕΠ μάλλον μειώνεται, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να μειώνεται χωρίς όμως να κινδυνεύουν τα κονδύλια προς τους στοχότερους ανθρώπους του κόσμου. 23.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα να σας θυμίσω. Ήταν 36.000 παιδιά κάθε μέρα. Κοιτάξτε πόσο πρόοδο έχουμε κάνει. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερη πρόοδο ακόμα λοιπόν. Να ε, μείνουμε λοιπόν στο ΑΕΠ. Στους επόμενους, ε, στις επόμενες γενιές, στην επόμενη γενιά, δύο δις ακόμα θα ζήσουν πάνω στην ε, γη. Θα υπάρξει μαζική μετανάστευση αν εμείς δεν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Γι' αυτό κάνω αυτή την έκκληση. Εντάξει, αν πρέπει να μειώσουμε τα ποσά, οκ. Αλλά όχι και το, ε, και το ε, Μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ο κύριος Στάσινη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως εισηγητής για δημοσιονομικά θέματα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στηρίζω σταθερά τις δραστηριότητε που, που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνουν τις διμερείς σχέσεις και βελτιώνουν την παγκόσμια σταθερότητα και αλληλεγγύη. Γι' αυτό και είμαι υπέρα της ε, χρηματοδότησης του, του, του της εμπορίας ε, και του ICI. Ε, και επίσης ε, θα ήθελα να, συμβάλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διεθνοποίηση των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης σε χώρες μεγάλης ανάπτυξης, βοήθεια σε εμπορικούς εταίρους στην νότια και ανατολική γειτονία μας, καθώς και πόρους για τους υπάρχοντες διαλόγους υψηλού επέδου με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και τις αναδυόμενες χώρες. Όλες αυτές τις δραστηριότητες αν εκτελούνται σωστά, θα, βελτιω... θα είναι πολύ ωφέλιμε για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία τον εισηγητή κύριο Λαβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Είναι ο κύριος Φιέλνερ που δεν, έχει, ε, δεν είναι στην αίθουσα όμως. Οπότε τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Σούλαντ εξ ονόματος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Μπουλόν. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ τον κύριο Λαβία για την ε, συνθετική του δουλειά, γιατί πιστεύω ότι η απασχόληση πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια στο να υπάρξει κοινωνική διακυβέρνηση, πράγμα που περνά μέσα από δράσεις που ευνοούν τη συνοχή και την ε, ε, σύγκληση. Ο προπολογισμό του 2013, και θα είναι ο τελευταίο του πολιετού πλαισίου που είναι υπό εξέλιξη, θα πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό των προγραμμάτων που είναι στο τέλο τη εκτέλεσή του. Αντίθετα, θα πρέπει να δώσει μια δυναμική ώστε να βοηθήσει του νέου να βρουν θέσει απασχόληση και να βοηθήσει τι ΜΜΕ, που είναι η πρώτη δημιουργή θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να περιορίσουμε ε, τι προσπάθειε που κάνουμε για την ε, καταπολέμηση τη ενεργεία. Το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και να ε, δοθούν νέοι προσανατολισμοί. Να δούμε πού λείπουν οι ε, υπάλληλοι και να ενισχύσουμε προγράμματα όπως το μικρό πέρες και μικροχρηματοδότησης. Γι' αυτό και οι δράσεις που γίνονται από τις μικρές, ε, μεσαίες ή και μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και από τις πολύ μεγάλες, θα πρέπει να στηριχθούν οικονομικά από την Ένωση. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος Επιτροπής Βιομηχανίας, ο κ. Μπουτικόφερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σαν πράσινος βουλευτής της Επιτροπής δεν συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους σχετικά με το πρόγραμμα ΙΤΕΡ και σαν εισηγητής της Επιτροπής ΙΤΡΕ πρέπει να σας πω ότι συμφωνούμε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους για την Ευρώπη του 2020 δηλαδή την ενεργειακή πολιτική που είναι ένα επίπεδο η έρευνα και η καινοτομία έχει προτεραιότητα και η στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως, ο κύριος Σταυρακάκης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται με την οικονομική και κοινωνική κρίση να βάζει σε δοκιμασία τους προϋπολογισμούς όλων των χωρών οι οποίοι καταρτίζονται στη βάση εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών. όσον αφορά την πολιτική συνοχή όλοι γνωρίζουμε κυρία πρόεδρε ότι είναι το κύριο και πιο κατάλληλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει την ευρωπαϊκή ένωση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. στο τέλο του 2011 είχαμε, μια, είχαμε ένα σημαντικό αριθμό καθυστερημένων πληρωμών που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσω τη διάθεση επαρκών πιστώσεων πληρωμών το 2012 οι ελλείψει στι πληρωμέ είναι πιθανό να επιδεινωθούν το 2013, όπου η εφαρμογή των προγραμμάτων τη πολιτική συνοχή παραμένει να επιταχυθεί. Γι' αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο θα πρέπει να προβούν στην άμεση ανάλυση και αξιολόγηση των ποσών και των αναγκών, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή των προγραμμάτων για το 2013. Εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αντιταχθούμε σε κάθε ενδεχόμενη μείωση του επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με τι ανάγκε αυτέ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο Επιτροπή Γεωργία, η κυρία Ντελάγκε. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο προπολογισμό για την Γεωργία αυξάνεται κατά 1,6. Αυτά είναι φραγκορίφραγκα σε σχέση με το 7% που στο παρελθόν πρέσβευε η Επιτροπή. Και Λοιπόν, στο για τα κρατημέλη ε, έχουμε τώρα τη στήριξη των εισοδημάτων και αυτό είναι μια, μια μια, μια, μια, μια, μια από τις αιτίες του ότι θα πρέπει στα παλαιότερα μέλη να σφίξουμε το ζωνάρι. Τι θα γίνει το 2013, τι θα γίνει με, τα, με τις τιμές. Υπάρχουν κάποια πολιτικά προγράμματα βέβαια. Θα πρέπει αυτά να τα προσέξουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι κοινωνικέ αγορέ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει καλύτερα να διαχειρίζεται τα πιλωτικά προγράμματα. Γιατί αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα στο, στο, στο παρελθόν. Επίση και η, η εποπτεία των τιμών είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για όλου. Δεν έκανε όσα θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει, να λάβει υπόψη ότι υπάρχει κρίση και χρειάζεται κάποιο είδου παρέμβαση γιατί και στα οποροκυπευτικά, φρούτα και εκεί θα πρέπει να κάνει περισσότερο. Ευχαριστώ. Πετροπή Λίμπε, ο κύριος Γιακολίνο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μια τόσο περίπλοκη εποχή όπου με δελτίο θα γίνονται οι δαπάνες θα πρέπει να έχουμε έναν λογικό προϋπολογισμό. Και η προσπάθεια του Τζοβάν Λαβία είναι ένα προφανές ε, μήνυμα για το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα και μπροστά σε τόσες δυσκολίες. Και εμείς ε, σημειώνουμε τις υποδείξεις ε, που λάβαμε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού και τις λάβαμε υπόψη ως θετικό μήνυμα αν στο Frontex στο θέμα που σχετίζεται με το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Ωστόσο, όταν ε, διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών και το 2013 που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αναφέρομαι ιδιαίτερω σε εκείνο τον κατάλογο πολιτικών προτεραιοτήτων όπου, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να μην αμφισβητηθεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κυρία Πρόεδρε. Εκεί μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, κάποια περισσότερα πράγματα και το ίδιο θα μπορούσαμε να, κάνουμε, να το λάβει υπόψη η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Συνταγματικές υποθέσεις, ο κύριος Γκερέρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Κύριε Επιτροπέ, εγώ ήμουν οσογητή στην ε, Συνταγματική Επιτροπή και επομένω, ε, ξέρετε, εδώ θέλαμε ε, ένα συνεπή προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόκειται για θετικό καταλήτη για κάποιε επενδύσει. Ακριβώ λοιπόν η περίοδο κρίση χρειάζεται να ακούγεται ενιαία φωνή όσον αφορά τον προπολογισμό από τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε απασχόληση και να δημιουργεί ανάπτυξη στι χώρε μα. Το 2013 είναι προεκλογική χρονιά. Και γι' αυτό και η Συνταγματική Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται, προβλέπεται μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση ενημέρωση των πολιτών. Να ξέρουν τι διακυβεύεται στι ευρωεκλογέ. Επίσης θα πρέπει να τους ε, ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη συμμετοχή στον πολιτικό βίο τη Ένωση. Οπότε, ακριβώ για αυτού του λόγου θα πρέπει να έχουμε ένα συνεπή συγκροτημένο προπολογισμό ούτω ώστε να μπορούμε ε, να βιονίσουμε τον πολίτη όλοι μαζί με φωνή. Επίση θα πρέπει να δούμε ε, το νομοθέτημα κοινοτόπιο το οποίο τον Απρίλιο τέθηκε σε ισχύ για κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίε κατέβηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε και θα χρειαστεί τελικά να γίνουν κάποιε ακροάσει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει επομένω και πλευρά προπολογισμού θα πρέπει να μπορούμε να καλύψουμε αυτέ τι ακροάσει για να γίνουν όπω πρέπει. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, η κυρία Χάνιμπολ δεν βρίσκεται στην αίθουσα, οπότε ξεκινάμε με τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ε, εξ ονόματος του ΕΛΚΟ, ο κύριος Λαμασούρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κρέμεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Την περασμένη Παρασκευή ομόφωνα ενέκρινε το Συμβούλιο ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη και αποφάσισε να δώσει για δύο χρόνια 55 δις στα διευθυντικά ταμεία επιπλέον για να χρηματοδοτήσει τα μελλοντικά σχέδια. Αυτή η πρόταση ήταν ευθύη, ρεαλιστική και λογική. Σέβεται το ανώτατο όριο δαπανών που είχε οριστεί πριν από πέντε χρόνια. Βασίζεται σε, βασικές, σε σημαντικές προσπάθειες που είχε κάνει η Κομισιόν, στην οποία ο φόρο τιμή και στις προσπάθειες που κάναμε για οικονομικά αποδοτικά προγράμματα αλλά έχει νόημα μόνο αν αυτές οι πιστώσεις που ανακοινώθηκαν μπορούν όντως να κινητοποιηθούν, άρα να δεσμευθούν και να καταβληθούν μέσα στο προπολογισμό του τρέχοντος έτους και στον προπολογισμό του 2013. Άρα λοιπόν τίθεται το εξή ερώτημα. Οι μόνιμοι εκπρόσωποι θα θάψουν από την επόμενη εβδομάδα και κλεισμένο το θηρόν την επίσημη απόφαση που έλαβαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων πριν από λίγε μέρε. Αν η Ένωση σήμερα στενεί οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν πια εμπιστοσύνη, οι, δημοσιο... οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, αμφιβάλλουν. Ε, αυτό οφείλεται στο ότι οι κυβερνήσεις αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα, μάλλον χρησιμοποιούν τα όργανα που τους περιβάλλουν για να λάβουν αποφάσεις αντιφατικές. Κανείς δεν καταλαβαίνει πια τι αποφάσεις λαμβάνονται. Όταν όμως καίγεται το σπίτι μας, τέτοιου είδους παιχνιδάκια δεν επιτρέπονται και θα είναι η ευθύνη της Κυπριακής Προεδρίας για την οποία να εκφράσω τη λύπη μου που αποουσιάζει για τις αποφάσεις που θα ληφθούν έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην φαίνει ως ένα, μια διάσκεψη κορυφής ανικανότητας ή υποκρισίας. Ευχαριστώ. Ξενόματος των Σοσιαλιστών, η κυρία Γκαρδιά Ζαμπάλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επίτροπε. Λέμε για το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο αφού στην περσινή εβδομάδα να εκταμιευθούν 120 δις. Δεν είναι αυτό φραγκοδίδι, φραγκά και τώρα το Συμβούλιο ε, προσέχει κυρίως την λιτότητα. Και εδώ το Μάρτιο τα ίδια είχαμε πει και είχαμε πει ότι κάνουν λάθος πολιτική, θα πρέπει να αλλάξουν ρότα και από ό,τι φαίνεται άρχισαν τα πράγματα να μεταστρέφονται στο Συμβούλιο και δεν προσέχουν μόνο αυτή την λιτότητα, το οποίο και αυτή χρειάζεται. Αλλά και επίσης μιλάνε και για δημιουργία ανάπτυξη ε, βιώσιμης, είναι σημαντικά τα 120 δις, αλλά επίσης έχουμε και ε, κάποια εργαλεία για τα οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε κάποιες επενδύσεις. Μιλούμε για τον κοινωτικό προϋπολογισμό, ο οποίος 151 ε, δις τα θέτει εις, ε, τη διάθεση κοινότητα. Δηλαδή περισσότερο από τα 120 δις τη πρώτης εβδομάδα. Θα πρέπει όμω οι Υπουργοί Οικονομικών να συνεχίσουν την ίδια ρότα που όπως είπε το Συμβούλιο την εβδομάδα και να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Επομένω και να εφαρμόσουν τι ίδιε αρχές στον προπολογισμό και σε αυτόν τον προπολογισμό για το 12 και για το 13 γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να, να υπάρξουν τα χρήματα του για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές και τις δεσμεύσεις μας. Τα είχαμε πει και είχαμε δίκιο. Σήμερα επομένω φτάσαμε να έχουμε το, κάποια προγράμματα όπω το 7ο για την ε, έρευνα, το οποίο μα έχουν παραλύσει η λήψη χρηματοδότηση. Γι' αυτό και ζητεί το Συμβούλιο ε, να δούμε τι θα γίνει και το είπαμε και εμεί στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να βρεθεί το χρήμα ούτω ώστε ε, να εκτελέσουμε αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν για να έκρινε τη συνάντηση κορυφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 έχει υποχρεώσεις ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου που καλύπτουν την ε, στρατηγική του 2020 για την Ευρώπη ε, και και αυξάνουν τις δεσμεύσεις 64 δισεκατομμύρια ιδίω αύξηση 3,5% για την βιώσιμη ανάπτυξη σχετικά με την ανάπτυξη ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την απασχόληση των νέων και προγράμματα ε, όπως ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα για να προωθήσουν την ανάπτυξη που είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη εάν κοιτάξουμε τους αριθμούς αυτούς ε, του προπολογισμού βλέπουμε ότι ενέρχονται υποχρεώσεις σε σύνολο 138 ε, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ και σε σχέση με το προηγούμενο έργο προηγούμενο έτος έχουμε μία σημαντική αύξηση για τις επενδύσεις που φτάνουν μέχρι και 12% για να προωθηθούν τα προγράμματα σε αυτό το χώρο. Όσον αφορά το σύνολο των πληρωμών έχουμε μία αύξηση 6% για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις δεσμεύσεις της τωρινής περίοδου με ε, τις υποχρεώσεις των προηγουμένων δημοσιονομικών περιόδων με ένα δύσκολο εγχείρημα διότι το 2013 για την ψηφιακή ατζέντα στην Ευρώπη θα χρειαστούμε την καλύτερη τεχνολογία και θα πρέπει να προωθήσουμε το μέτρο αυτό. Είναι άλλωστε μία, ένα ένασμα το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε από κοινού με το Συμβούλιο διότι έτσι θα μπορέσουμε ε, να έχουμε περισσότερες οικονομίες αν οι συζητήσεις αυτές γίνονται στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τους πράσινους τώρα, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Τρίπολη ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο σήμερα το πρωί μας είπε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι το αποφασιστικό μέτρο για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Συμφωνώ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι σαν επίτροπος το επανέλευε και αυτό που δεν δέχομαι τώρα είναι να τονίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε είναι μέρος της κοινοτικής μεθόδου. Πρέπει να συζητάμε με το Συμβούλιο και μόνο μετά υπάρχει ένας ενιαίος προϋπολογισμός μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Πρέπει τώρα να κοινοτοποιήσουμε όμως γρήγορα 55 δισεκατομμύρια για να δημιουργήσουμε ενάψματα αναπτυξιακά στην παιδεία, στην έρευνα, στη βιώσιμη ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλους πολύ καλούς στόχους. Το Συμβούλιο όμως παρέλειψε να μας πει από πού θα βρει αυτά τα χρήματα βραχυπρόθεσμα. Και γι' αυτό στηρίζω αυτά που ελέγχθησαν μόλις, ότι το Συμβούλιο είναι σχιζοφρενές πολιτικά. Από τη μια μεριά θέλει να κάνει αυξήσεις και από την άλλη πλευρά δεν είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει ούτε το 2012 ούτε το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις δηλώσεις των κρατών μελών ήταν επιφυλακτική. Ε, τονίζει όμως ότι πρέπει να σεβαστούμε τις συνθήκες, γι' αυτό και εμείς απαιτούμε απαιτούμε από το Συμβούλιο και την Κυπριακή Προεδρία να είναι θαραλέα, να είναι Ευρωπαίοι και να φροντίσουν να κινητοποιηθούν οι πληρωμές διότι διαφορετικά θα απογοητεύσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη με αυτό το οποίο αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εξ του ΕΛΚΑ, ε, κύριος το ECR, με συγχωρείτε, ο κύριος για δύο λεπτά. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις σαν προηγουμένου. Διακυβεύεται η ικανότητά μας να συμβαδίσουμε με τον υπόλοιπο κόσμο, πράγμα που θα καθορίσει το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Ο προϋπολογισμός θα είναι το κλειδί για αυτό το μέλλον και ότι η πιο πιεστική προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ώστε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη βασιζόμενη σε πλήρως λειτουργούσα ενιαία αγορά και μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων που δαπανώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη, επενδύσει ε, στις υποδομ... συνοριακές υποδομές και επενδύσει ε, σε... στην ευρυζωνική σύνδεση. Αυτά όλα σημαίνουν επενδύσει στην πραγματική ζωή και στο μέλλον. Αλλά σημαίνουν επίσης ότι σε έναν αυστηρά περιορισμένο προπολογισμό θα πρέπει να μπορούμε να δαπανίσουμε εκεί μόνο όπου υπάρχει πραγματική ε, απόδοση των χρημάτων που επενδύουμε θα έπρεπε να ξανακοιτάξουμε τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς τομείς δαπανών. Θα πρέπει να θέσουμε δύσκολα ερωτήματα. Για παράδειγμα, οι περασμένες επενδύσεις σε προγράμματα διευθυντικά έφεραν τα, απέφεραν τα ωφέλη που έπρεπε. οι προτάσεις μεταρρύθμισης για την κοινή κυριακή πολιτική πραγματικά θα αποδώσουν μετρήσιμα περιβαλλοντικά ωφέλη και με ποιο κόστος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Το το των ε, οικονομικών αυτών προκλήσεων, αυτός ο προπολογισμό χάνει την ευκαιρία να αναζητήσει αυτές τις νέες προσεγγίσεις. Αντίθετα, μια από τα ίδια μας προτείνει. Τις ίδιες πολιτικές με περισσότερα στα Πρόεδρε, ε, το σώμα μας θα έκανε λάθος αν θεωρούσε πως μπορεί να συνεχίσει αυξάνοντας τις δαπάνες τη στιγμή που οι λαοί της Ευρώπης ε, βιώνουν τις περικοπές και τη λιτότητα. Θα έπρεπε να παγώσει το μέγεθος του προϋπολογισμού κανονικά. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Γκουε, η κυρία Σόζα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Ευρώπη η μοναδική απάντηση των κυβερνήσεων στις ανάγκες των πολλαών ήταν η λιτότητα. Ε, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη αλληλεγγύης, όχι αυτή την Ευρώπη της τιμωρίας. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο με την δημοκρατική νομιμότητα άμεση. Δεν μπορεί να παραδίδει στις κυβερνήσεις την αποκλειστικότητα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ήδη γνωρίζουμε ποια είναι η συνταγή. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσουμε κατά της εντολής. Ε, έχουμε πολλές και βαθιές αποκλήσεις ε, με το μεγλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου. Δεν θα στηρίξουμε, για παράδειγμα, τις άμεσες μεταφορές για τις ε, πολυεθνικές ε, των φαρμάκων, ούτε τις επενδύσεις για τη δημιουργία μιας Ευρώπης οχυρού. Αντίθετα θα υπερψηφίσουμε ε, τα προγράμματα υπέρ της ανάπτυξης ώστε να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση στην κρίση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για υποχρεώσεις που ήδη έχουν αναλυφθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Οι βασικοί παραλήπτες δεν είναι παρά η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Με λιγότερους πόρους θα έχουμε απλώς λιγότερη απασχόληση, περισσότερη φτώχεια και μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν είναι τώρα ο καιρό για μισόλογα, ούτε για μισές αποφάσεις από πλευρά των ηγετών της Ευρώπης. που μέχρι τώρα ακολουθούν τις αγορές και τις τράπεζες θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Να ε, τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε εδώ και εκεί έξω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, της ομάδας ε, D, η FD, η κυρία Ανδρέασεν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να και πάλι τα ίδια. Μέσα στη χειρότερη κρίση που θυμάται ο κόσμος, εδώ πέρα μας προκύπτει κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ρεαλιστικό και οίκιστα υπεύθυνο, γιατί θα πρέπει να ε, δούμε το πώς είναι δυνατόν η... να ζητεί εδώ πρέπει ψηφία μία αύξηση του 6,8%. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι είναι μία αυθεντική ανάπτυξη που μπορεί ο προπολογισμό να κινητοποιήσει έτσι. Αυτό είναι απλά γελίο γιατί έχουμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων τα οποία έχουν, έχουν, έχουν, έχουν πάει στο πηγάδι αυτό χωρίς πάτο και δεν φέφεραν καμία ανάπτυξη. Πολλοί από μας πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιε πολιτικές ε, τι τις ευθύνες της σχετικά με την κρίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίω έχει αποτύχει όσον αφορά τον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων και νομίζω ότι αυτό μα το πιστεύτηκαν οι φορολογούμενοι. Να έχουμε κάποια στοχευμένα, στοχευμένους πόρους σύμφωνα με την νομοθεσία ε, και να έχουμε συνολικά κάποιο όραμα και τελικά εμεί αποτύχαμε ναι, κύριε Κάμερον ναι, το μήνυμα με ακούτε είναι για σας συνεχίστε να στέλνετε λεφτά στις Βρυξέλλες αν το κάνετε αυτό, τότε διαβιβάζετε εξουσίες σε μια γραφειοκρατία η οποία είναι ανεύθυνη, η οποία είναι σπάταλη, οπότε ε, λυπηθείτε τους ε, Άγγλους και κόψτε, κόψτε τις εισφορές σας στον, στο, στον κορβανά της ε, Ένωσης και απαιτήστε πάγωμα των δαπανών. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ έχουμε μία ε, μεγάλη διαρθρωτική κρίση στην Ευρώπη η οποία οδηγεί σε μεγάλη ενεργεία των νέων. Είναι μία εκρηκτική κοινωνική ουσία η οποία ε, ταλαιπωρεί ε, ολόκληρες γενιές ανθρώπων και ζητά μία γρήγορη πολιτική αντίδραση. Επί αυτής της βάσεως ο προπολογισμό του 2013 είναι η σωστή αντίδραση του Κοινοβουλίου όπου υπήρξαν πολλές περικοπές ακόμη και στο προσωπικό των θεσμικών ογράμμων κατά τρόπον ώστε σε όλα τα επίπεδα να μπορέσει να εστιαστεί το ενδιαφέρον ή εις το μέλλον των νέων και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και να δημιουργήσουμε νέες προπτικές για τους νέους και για το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα οι υπόλοιποι ομιλητέ. Ξεκινάμε με τον κύριο Σούριαν για ε, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τον εισηγητή που είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο, όπως το ακούσατε. Ο προηγούμενο του 2013 θα πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της Ευρώπης. Νομίζω ότι περισσότεροι εξημών συμφωνούμε ότι βασική προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης, ε, η συρρήγνωση της παραγωγής. Πολλοί κατηγορούν τις τράπεζες. Κατηγορούν την περικοπή των χορηγήσεων και δανείων. Και επίσης την έλλειψη εξυγίανσης στον τραπεζικό τομέα. Η κρίση μας έχει στριμώξει σε ένα διέξοδο από το οποίο πρέπει να βρούμε την λύση, την έξοδο, όμως το να κάνουμε τέτοιου είδου ε, προϋπολογισμό ε, θα πρέπει να δούμε πώς με αυτόν τον προϋπολογισμό τέλος πάντων θα βρούμε ανάπτυξη και απασχόληση. Όμως, να μην κολλάμε και να θέλουμε να συνεχιστούν τα προγράμματα όπως ήταν πριν την κρίση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τον προπολογισμό τη χρήση του 2013. Θα πρέπει να δείξουμε τόλμη και θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μα σε προγράμματα που βοηθάνε απασχόληση και ανάπτυξη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να αποκρίνεται ταχύτερα όσον αφορά τα, τα όσα θέτουν τα κράτη-μέλη. Έτσι θα έχουμε επιτυχή διαχείριση τη κρίση. Εάν συνεχίσουμε να, να, να, ονειρευόμαστε για μία απορροφημένα ε, κεφάλαια πόρου, δεν κάνουμε τίποτα. δεν θα κάνουμε τίποτα καλύτερο. Να σταματήσει αυτός ο μύθος των μη απορροφηθέντων κονδυλίων. Οι πιστώσεις πληρωμών πρόκειται να αυξηθούν. Εμείς θα πρέπει επίσης να τρίσουμε τις δεσμεύσεις μας. Θα πρέπει τα προγράμματα να προεκοδοτηθούν. Επομένω, εγώ είμαι θετικός. Σας ευχαριστώ. κύριος Βόν για 1,5 λεπτό.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 Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λαδία για την εξαιρετική του έκθεση. Εγώ παίρνω το λόγο ως εισηγητή για τα άλλα τμήματα υπό την κατηγορία 5 και ίσω δύο λόγια για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται την επιστολή από τον Επίτροπο που καλούσε όλα τα θεσμικά όργανα να μείνουν κάτω από το 1,9% όσον αφορά την αύξηση για το επόμενο, τον επόμενο έτο. και εμεί είπαμε στι εκτιμήσει μα ότι είχαμε στόχο αύξηση 1,9 αυτή τη στιγμή για την ώρα. Γιατί αυτό που κάναμε στο Κοινοβούλιο να φτιάξουμε μια ομάδα εργασία που θα εξέταζε τι εξοικονομήσει στο Κοινοβούλιο. Εξετάζουμε ας πούμε, το κόστος των οδηπορικών και για το μέλ και για το προσωπικό και Βλέπουμε και μελέτες από τα κράτη-μέλη και από το Αμερικανικό Κογκρόσο. Γύρω στο Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποιες εξοικονομήσεις στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε έτοιμη και ολόκληρη έκθεση. Να πω δύο λόγια για τον προπολογισμό των άλλων θεσμικών οργάνων. Η Κομισιόν αρχικά πρότεινε μια αύξηση 3,2%. Από ό,τι κατάλαβα το Συμβούλιο θα προτείνει αύξηση 1,8%. Πράγμα βέβαια που είναι πολύ κοντά στο 1,9% που αρχικά πρότεινε η Κομισιόν. Αν και πιστεύω πως πρέπει να εξετάσουμε όλα τα θεσμικά όργανα μεμονωμένα. Ξέρουμε για παράδειγμα το Δικαστήριο και η Εξωτερική Υπηρεσία ε, ήδη λένε πως θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερη αύξηση, αλλά εν γέννη θα πρέπει να στοχεύσουμε σε μια αύξηση 1,9% αν όχι και λιγότερο και μπορούμε να πούμε ότι ως Κοινοβούλιο και οι υπόλοιποι να πούν ότι έχουμε μια πραγματική περικοπή στο διοικητικό κόστος των θεσμικών μας οργάνων. Θα ήταν πολύ θετικό για το Κοινοβούλιο και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Grazie. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φάιμον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν κάθε χρόνο συζητάμε για την εντολή, για τον τριμερή διάλογο, για τον προϋπολογισμό και για τον, ε, τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Θέλω όμως να ζητήσω κατανόηση. Έχουμε προσπαθήσει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να ε, ζητά πράγματα ανέφικτα. Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκη και δεν θα βελτιωθεί του χρόνου. Οπότε δεν είναι δυνατόν τα κράτη μελη να μας επιβάλλουν ε, αυξήσεις στον προϋπολογισμό. Πρέπει να προσπαθήσουμε ο προϋπολογισμός για του χρόνου να μπορέσει να γίνει αποδεκτός εγκαίρος για να μην έχουμε καθυστερήσεις και να μην χρειαστεί να λειτουργούμε με προσωρινά μέτρα. Οποιαδήποτε διένεξη για μικροθέματα θα έθετε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο και αυτό δεν πρέπει να το επιτύχουμε διότι του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτύχει σωστές αμοιβέ ε, για τις άμεσες πληρωμές προς τους νέους γεωργούς στα νέα κράτη-μέλη και ελπίζω θα μπορέσει να το πραγματοποιήσει. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Βουλόσοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο είχαμε κρίνει ότι ανάμεσα στις προτεραιότητες ε, για το Κοινοβούλιο ήταν η στήριξη της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη στρατηγική 2020, είμαι τη ίδια άποψης όσον αφορά τη στήριξη προς τις ε, μικρομεσαίες και του νέους. Το σχέδιο που υποβάλλει η Κομισιόν προχωρεί προς αυτή την κατεύθυνση και είναι άρα ικανοποιητικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κοινοτικός προπολογισμό είναι ένα μέσο πραγματικών επενδύσεων πολύ ισχυρό το οποίο χρειαζόμαστε για να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης σε όλα τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό και στηρίζω το σχέδιο της Κομισιόν σε σύγκριση με τις άλλες προτάσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό που με δυσαρεστεί είναι η μείωση των, των πιστώσεων για το, σχέδιο, για το πρόγραμμα Progress που έχει στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ε, εάν προβλέπουμε να δώσουμε στους νέους εργαλεία για την ανάπτυξή τους, για να βρουν θέση απασχόλησης, αυτό θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε την κρίση. Δεν πρέπει να δίνουμε ψάρια σε αυτούς που πεινούν, αλλά να τους δώσουμε ένα καλάμι ψαρέματος. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Άρτογκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγα και είδα μια ταινία, τη τέταρτη εκδοχή του Ice Age. Και όταν ερωτήθηκε με χώρα γιατί έχει τόσα πολλά προβλήματα, απάντησε ότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε ανόητοι, γι' αυτό έχουμε τόσα προβλήματα. Ίσως ε, αυτή είναι η απάντηση και για τη συζήτηση που έχουμε για την εντολή για τον προπολογισμό το 2013 και αν δούμε την πρόταση για 6,8 αύξηση του προϋπολογισμού και δούμε και τον κατάλογο των προτεραιοτήτων, θα λέγαμε ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2013 τι θα αυξηθεί και τι θα γίνει τα πάντα και τι δεν αυξάνεται. Ξέρουμε εμείς οι πολίτες πώς έφτασε η Ευρώπη σε αυτά τα ε, προβλήματα. Ποιος φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μα είναι ε, δυνατόν είναι τόσο ανόητη. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, la parola all'onorevole per due minuti. Κυρία Γεντζεγεύσκα, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική έκφαση της αλληλεγγύης μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαλείο που δεν εξυπηρετεί μόνο την εξίσωση των διαφορών στην ευημερία μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, αλλά κυρίω ενισχύει τι επενδύσει, την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί νέε θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, έχουμε πολλέ ιδέε για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ήδη πολλά εργαλεία και μηχανισμοί. Αρκεί να αλλάξουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, το πρόγραμμα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και το πρόγραμμα για τη διαβίου κατάρτιση. Και η υλοποίησή τους δεν εξυπηρετεί μόνο τους άμεσου οφειλέτες, αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τι προκλήσει του 21ου αιώνα, κυρίως ε, την ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, σημαντικό επίπεδο δαπανών στον προπολογισμό του επόμενου έτους, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις ε, ενηλυμένε μας υποχρεώσεις και τις υποσχέσεις και να μπορέσουμε να διέλθουμε από την ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την ευάθυνση των διαφορών σε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο και τις δαπάνες ε, των διαφόρων τμήματων του προϋπολογισμού γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις υποχρεώσεις μας. Γιατί η αύξηση των πληρωμών 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 2012, είναι η ελάχιστη αύξηση που θα έπρεπε να δεχτούν και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα θέματα διάσωσης και στα τρέχοντα προβλήματα και στις ε, άμεσες λύσεις. Θα πρέπει να έχουμε και μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μακρόπορη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Τζοκ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Συζητούμε εδώ την ανταγωνιστικότητα και θα ήθελα να τονίσω ότι το έτος 2013 είναι το τελευταίο έτος του παρόντος προγράμματος ε, πλαισίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε με φιδό τα κονδύλια ε, και να πιάσουν τόπο και θα χαιρόμουν να αυξηθεί η πυρκοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μην μειωθεί και να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης θα χαιρόμουν τα ομόλογα έργου να γίνουν ένα πείραμα που να στεφτεί με επιτυχία και τα προγράμματα υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα έργα. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω κύριε Επίτροπε ότι καλωσορίζουμε το πρόγραμμα ITER μεν, αλλά το επιπλέον κόστος του προγράμματος αυτού θα πρέπει να εξασφαλιστούν από άλλες πηγές. Δηλαδή να μην ε, είναι εις βάρος άλλων προγραμμάτων. Βλέπε έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Να μην χαθούν από εκεί τα χρήματα και να βρεθεί μια λύση όπως βρέθηκε και φέτος άλλωστε. Επίσης θα έλεγα ότι Υπάρχει και ένα πρόγραμμα που δεν έχει ε, τη σωστή ε, επιδότηση, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, δεν είναι τώρα του παρόντος. Ευχαριστώ. Τερό για ένα λεπτό. Κύριε rouva Πουχεμίες. Hyvä komissaari, raportööri ja kollegat. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, Κυρίες και κύριοι, ο, πρόεδρο, ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι δύσκολο. Ζητάμε τεράστιες θυσίες από τα κράτη-μέλη και από τις ε, κεντρικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, υγείας κτλ. Σε μια τέτοια στιγμή δεν μπορούμε να μένουμε κλεισμένοι στους πύργους μας και να μην γνωρίζουμε ποια είναι η καθημερινή κατάσταση των πολιτών το, η, ε, το πάγωμα των πιστώσεων σε διάφορους τομείς επίσης μας αφορά. Αν θέλουμε μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού κινδυνεύουμε να βλάψουμε το όνομά μας και να θεωρηθούμε αδιάφοροι. Στην έκθεση πρέπει να επιδιώξουμε να αποφύγουμε τις άχρηστες δαπάνες, τις σπατάλες. Δεν θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματα που μπορούν να κάνουν από μόνο τους τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χολμάγερ, παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των ε, οργανισμών ε, agencies. Το έτος 2013 αλλά και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 14 με 20 δεν έχουν συγκεκριμένη στόχευση στη χρηματοδότηση. Παράδειγμα, έχουμε ε, νέους ε, οργανισμούς εποπτείας εάν ε, πραγματικά θα πρέπει να ανταποκριθούν στο έργο τους και στην εντολή τους που ξανασυζητήσαμε και το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ανάλογα για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα καθήκοντα. Αλλιώς όλο το σχεδιασμό που έχουμε κάνει δεν μπορούμε να τον εφαρμόσουμε. Δεύτερο παράδειγμα, Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ έχει πάρα πολύ χρηστή οικονομική διαχείριση. Το έτος 2011 έχει και μεγάλες μεταφορές πιστώσεων γιατί άρχισαν αργότερα τα προγράμματα. Και ε, τώρα τιμωρούν μείον 10% και ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσει και ένα νέο κέντρο για την πάταξη του κυβερνοεγκλήματος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι λογική η χρηματοδότηση των οργανισμών και ε, ταυτόχρονα να ε, αληθέψουμε τη λειτουργία του διοικητικών του συμβουλίου για να δούμε πώς ε, μεταφράζεται αυτό στην πράξη και πώς λειτουργούν πραγματικά οι οργανισμοί αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Φερνάντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνεται για το 2013 έχει προ... Ε, προβλέπει ενίσχυση 6,8% σε σχέση με τον προπολογισμό του 2012 σε ό,τι αφορά τι ε, πιστώσει πληρωμών, που φτάνουν έτσι στα 138 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ευελπιστώ ότι η αύξηση αυτή που προτείνουμε να σταθεί επαρκή για να αντιμετωπίσει τι ήδη υποχρεώσεις υποχρεώσει Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων τις επενδύσεις που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι στα τέλη του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να επιστρέψει περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν οφειλόμενα και ε, κυρίως ε, από πληρωμές που απαιτούνταν και εξαιτία του χαμηλού επίπεδου των ε, κονδυλίων που είχε. Αυτό ε, εξηγήθηκε από την αδιάλακτη στάση του Συμβουλίου που έσκαψε μόνο το λάκκο του. Και δεν θα έπρεπε να εμποδιστούν ε, οι πληρωμές των ε, υποχρεώσεων που ήδη είχαν αναλυθεί και που ήταν σημαντικές για να εξασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και ταυτόχρονα να υλοποιήσουν την, οικονομική, οικονομική και, την κοινωνική, οικονομική και ταφική συνοχή. Δεν θα πρέπει αυτή τη φορά να, να δημιουργήσουμε προσκόμματα στην στην αύξηση αυτών των, της πληρωμής, ε, των επιστώσεων πληρωμών. Νομίζω ότι ε, με τις προτάσεις αυτές ε, θα δώσουμε έμφαση στην ευφυή ανάπτυξη που θα περικλεί και δεν θα αποκλεί κανέναν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προπολογισμού του 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Ματέρα στην του, eh, Οπότε θα δώσω ε, το λόγο στους υπολείπους στο Catch Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να είναι μηχανισμός ε, αλληλεγγύης ε, και επενδύσεων. Γι' αυτό και η μείωση των ε, πληρωμών για την υλοποίηση των πολιτικών ε, και μάλιστα πολιτικών ανάπτυξη και απασχόληση θα είναι επιβλαβή σε μια τέτοια μείωση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης και πολλές χώρες μέλη το 2012 χρειάστηκαν ακριβώς για να καταπολεμήσουν την κρίση να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό τους. Είναι ανησυχητικό ότι σε ό,τι αφορά τα ραλ, τα υπόλοιπα προς καθάριση, υπάρχει πρόταση μείωσης ε, των πληρωμών. Και μάλιστα ε, θα έχουμε συσσόρευση πληρωμών για το 2013. Θα χρειαστούν πολύ περισσότερα κονδύλια. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τα ράλα, αλλιώ θα έχουμε δημοσιονομικέ δυσκολίε. Ο περιορισμό των πιστώσεων πληρωμών θα διακυβεύσει την ίδια την πολιτική συνοχή, που θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην αναζωγόνηση τη οικονομία και την επαναφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ανάπτυξη οικονομική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Βασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά στοιχεία εσωτερικής πολιτικής, ανάπτυξης, ε, απασχόλησης όταν καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό. Εγώ είμαι υπέρ της αύξησης ε, των κονδυλίων που δεσμεύονται υπέρ των νέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά είναι, ξέρετε, μικρομεσαίες, αλλά προσελκύουν ε, μόνο πολύ χαμηλό ποσοστό των συνολικών επενδύσεων. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα στις μικρομεσαίες αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση με επιτυχία. Η οικονομική λογοδοσία, θυμίζω, είναι πάρα πολύ σημαντική και τώρα σε τους καιρούς δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και ο προλογισμός της Ένωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις πολιτικές ανάκαμψεις των κρατών μελών, έτσι ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ λίγο να συμβάλλω στη συζήτηση. Βρισκόμαστε στο τέλος τώρα της επτά τους προγραμματικής περίοδου και αντιμετωπίζουμε διάφορες πληρωμές που πρέπει ε, να δώσουμε ε, για τη συνοχή ας πούμε και από προηγούμενα έτη. Μα είναι τρελό. Τα πρώτα χρόνια επιστρέφουν τα χρήματα στα κράτη-μέλη, στους καθαρούς συνεισφορείς. Και τα τελευταία χρόνια αρνούνται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ε, πρώτα τους δώσαμε πίσω τα λεφτά και τώρα είναι λογαριασμοί και δεν μπορούν να τους καλύψουν. Μα τι θα γίνει, κάθε χρόνο συμμαζεύουμε ε, αυτά που περισσεύουν, τα δίνουμε στα κράτη-μέλη και όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού δεν έχουμε χρήματα. Τι να κάνουμε, δεν, δεν μπορούμε λίγο να βάλουμε μια τάξη σε αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει περίπλοκη και θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό. Είμαι όμως πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν θα πρέπει να έχει υπερβολική συμμετοχή ε, στο αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης, τα κράτη-μέλη όλο και περισσότερο καλούνται να κάνουν οικονομίες και περικοπές. Και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να σεβαστούν την άποψη του Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη επίσης. Υπάρχουν αποθεματικά, ε, υπάρχουν ε, κάποια χρήματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν με σωστό τρόπο κάποιες πολιτικές. Παράδειγμα, έχουμε ένα σωρό λεφτά που δίνουμε στον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μπορεί να αξιοποιηθούν καλύτερα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Λεβαντόσκη. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι πλέον ε, πολύ της μόδας η σύγκριση των εθνικών προϋπολογισμών με τον ε, ευρωπαϊκό. Αυτό είναι μόνο εν μέρη δικαιολογημένο γιατί δεν υπάρχουν απόλυτες ομοιότητες ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πάντοτε είναι ισοσκελισμένος. Δεν υπάρχουν χρέη και ελλείμματα λόγω του μεγέθους. Είναι το 1% του ε, αλλά δεν Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο ποσοστό για να στηριχθούν τα θεσμικά όργανα. Και αυτό δεν έχει σχέση με τα 3 εκατομμυρία. Εν πάση περιπτώσει όμως μπορεί αυτό να δείξει ένα μέρος της λύσης για το πώς να ενισχυθούν η ανάπτυξη και οι ευκαιρίες για ε, θέσεις εργασίας. Πρέπει επίσης κάνουμε προσπάθεια να ε, εξοικονομήσουμε αυτά τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν και αυτή είναι μια ομοιότητα. Για πρώτη φορά από το, μέχρι το 2014 θα αρχίσει μείωση του προσωπικού, όχι αύξηση και αυτό αφορά δυστυχώ και του ε, οργανισμού στα γερμανικά και το λέω στην αγαπητή κυρία Χόλμα. Οι εξαιρέσει δεν κάνουμε. Εάν γίνουν εξοικονομήσει ε, επιδόσεων, αν χρειαζόμαστε ας πούμε προσαρμογή στα αναπτυξιακά μέσα συνεργασίας, ε, στην Λατινική Αμερική και την Ασία όπου κάποια προγράμματα δεν είναι αποδοτικά κάνουμε οικονομίες και αυτό φαίνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014. Αυτή τη στιγμή από όψη δαπανών βρισκόμαστε με 66 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από ό,τι είχαν συμφωνηθεί για την δημοσιονομική προοπτική 2007-2014. Αυτό είναι το καθαρό αποτέλεσμα των ε, εξοικονομήσεων των επιδόσεων και επίσης το, της αυστηρότητας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι όμως ο προϋπολογισμός είναι τα μέσα για την κάλυψη των δικαιολογημένων πληρωμών που οφείλονται σε εγκεκριμένα έργα στα κράτη-μέλη. Το 94% του προϋπολογισμού βγαίνει έξω από τις Βρυξέλλες. Το 6% αφορά τη διοίκηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν καθυστερούμε την πληρωμή, όταν δεν πληρώνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα των, επιστρο... των... πληρωμών προς τα ε, Υπουργεία Οικονομικών που ε, επιδεινώνουν την κατάσταση ρευτότητα στα κράτη-μέλη ή περιορίζει τις ευκαιρίες επενδύσεων στα κράτη-μέλη και δεν προσφέρει τα μέσα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα βουνό απλήρωτων υποχρεώσεων μελλοντικών λογαριασμών. Αυτό δεν είναι λύση. Ο προπολογισμό του 2014 είναι θέλω να πω ότι είναι λίγο σχιζοφρενικό να στέλνουμε τους λογαριασμούς στις Βρυξέλλες και μετά να γίνεται προσπάθεια να, γίνονται, να τηρούνται οι υποχρεώσεις. Ε, είναι δύσκολο. Ε, νομίζω ότι το 2000, ο προϋπολογισμός του 2013 δεν θα εκπλήξει ε, κανέναν ότι υπάρχουν ότι έχει ευξημένες, ε, ευξημένα αιτήματα πληρωμών. Μιλάμε για την αναψυξιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως ε, έχει και δημοσιονομικό σκέλος. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Λαβία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι φάνηκε, αναδύθηκε μεγάλη ε, πλειονότητα των τοποθετήσεων υπέρ της υποστήριξης της θέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είναι σαφές ότι οι ανάγκες πληρωμών θα πρέπει βεβαίως να ακολουθούν τις ε, δεσμεύσεις και την ανάληψη υποχρεώσεων προηγουμένων ετών. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι ε, σήμερα που έχουμε ένα ραλ που ξεπερνάει τα 207 εκατομμύρια ευρώ, ε, έχουμε επίσης και ένα τεράστιο όγκο πληρωμών ε, και οι λογαριασμοί είναι θεμητοί ακριβώς γιατί η ανάληψη υποχρεώσεων των προηγουμένων ετών ήταν ε, θεμητή και τώρα θα πρέπει να τιμηθούν αυτές οι υποχρεώσεις και η ανάγκη πληρωμών έχουν να κάνει περισσότερο με τους τίτλους που έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, με γέθεση της οικονομίας. Η μάχη λοιπόν για τις πληρωμές πρέπει να δοθεί και το Κοινοβούλιο με αυτή την εντολή για το τριμερή διάλογο δίνει ε, σημαντική ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητήσαμε διοργανική συνεργασία. Γιατί τη ζητήσαμε. Διότι είναι προφανές ότι χωρίς ε, μια κοινή αφετηρία ε, για τις πληροφορίες ε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μπορεί να καταλήξουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το είδαμε και πέρσι στη συνδιαλλαγή. Ε, κινήσαμε από διαφορετικές εκτιμήσεις. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις πληρωμές και σήμερα ζητούμε και με την εντολή μας το τριμερή διάλογο, ζητούμε από το Συμβούλιο να συμμετέχει και εκείνο στο διοργανικό διάλογο, γιατί μπορεί στο τέλος της αντιπαράθεσης, όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού για το 2013 να τελειώσουμε, ε, να κλείσουμε την υπόθεση του προϋπολογισμού, ε, τότε θα βρούμε τις πραγματικές ανάγκες μπροστά μας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι για την ειλικρινή συνεργασία και ελπίζω αύριο να με υποστηρίξετε για το τριμερή διάλογο και ελπίζω να περάσει αυτό με μεγάλη πλειοψηφία και να δώσουμε διαπραγματευτική ισχύ ε, στη συζήτηση που θα έχουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Τέλος της συζήτησης. Όπως είπατε και εσείς, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30.